Ladies and gentlemen, can we start? Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι. Okay. Λαμπρά. Ξεκινάμε. Σημείο 1. Υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης παρακαλώ. Έχουν επέλθει εξή αλλαγέ στη βασική ημερήσια διάταξη. Το 8 όσον αφορά την όσον αφορά τον κώδικα της Ένωσης για τις Βίζες έχει αναβληθεί. Το σημείο 8 παρακαλώ. Επίσης το σημείο 10 της κυρίας Κρυμάλη όσον αφορά την εξέταση για την εφαρμογή ορισμένων διεθνώς ε, standards προδιαγραφών σύμφωνα με τον κανονισμό και αυτό έχει αναβληθεί. Όσον αφορά την πρόταση που έρχεται εκ μέρους της αριστεράς που αφορά τη νομική βάση το θέμα της νομικής βάσης καθώς έχουμε ένα το τον Αλέξη Φόσφορο σαν ανησυχητή θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την νομική υπηρεσία και προτείνω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε και αυτό το σημείο για την επόμενη συνεδρία μας ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι παρακαλώ Κύριος Χρυσόβουλος παρακαλώ έχει το δρόμο ε, προτείνω να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη των εργασιών της Επιτροπής μας και να συζητήσουμε σήμερα κατά προτεραιότητα το θέμα της ισχύω του κανονισμού 833 του 2014 του Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία προκειμένου η Επιτροπή μας να λάβει απόφαση να εισηγηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα συνεδριάσει στις 15 έως 18 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο τη λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του Κοινοβουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του κανονισμού αυτού. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν επιδέχεται καμία αναβολή, διότι δεν υπάρχει άλλη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου έως τις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε λίγη η προθεσμία των 60 ημερών εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του κανονισμού αυτού και βέβαια πρέπει να επισημάνω ότι είχα εγκαίρως ενημερώσει με γραπτό μου σημείωμα στις 22 Αυγούστου όλα τα μέλη της Επιτροπής για την πρόθεσή μου να υποβάλω την πρόταση αυτή. Συνεπώς θεωρώ ότι το θέμα είναι απολύτως όριμο προς συζήτηση είναι ένα θέμα κέρια σημασίας όχι μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά γενικότερα για τη λειτουργία της Ένωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ένωσης σήμερα είναι το δημοκρατικό της έλλειμμα. Εδώ έχουμε μια απόφαση η οποία δυνητικά θα μπορούσε να πυροδοτήσει την επανέναρξη ενός ιδιότυπου ψυχρού πολέμου μεταξύ της Ένωσης και του μεγαλύτερου σε πληθυσμό και έκταση ευρωπαϊκού κράτους, δηλαδή της Ρωσίας, και η οποία ελήφθη χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοβουλευτική διαδικασία, διότι η ορθή νομική βάση ήταν και είναι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ο κανονισμός αυτός προβλέπει απαγόρευση εξαγωγών και όχι το άρθρο... Τελειώνω, τελειώνω. Και όχι το άρθρο 215 το οποίο προβλέπει μόνο χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Δεν αφορά μόνο χρηματοπιστωτικά ζητήματα ο κανονισμός αυτός. Λυπάμαι κύριε. Λυπάμαι. Σήμερα. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ο, Ιταλ... ο Ιταλός Υπουργός αναμένει ε, ε πρώτον πυλών ότι υπάρχει μία Στις 23-24 του μηνός Οκτωβρίου μπορεί να επιληθεί το θέμα αυτό και νομίζω πως υπάρχει αρκετός χρόνος για αυτό το θέμα. Πόσο μάλλον που αυτή, αυτό το θέμα αποφασίστηκε και κλεισμένο το θυρών στις συναντήσεις και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχουν λοιπόν τρεις λόγοι για την αναβολή αυτού του θέματος στην επόμενη συνάντηση. Υπάρχει συνένεση για την αναβολή. Βλέπω. Ενάντια ενάντια στην ψήφο. Για να είμαι ευγενής, επιτρέψτε με να πω κάτι. Να καθιστορήσω τον Ιταλό Υπουργό Ορλάντο. Εξοχότατε, καλωσορίσατε στην Νομική Επιτροπή και σας ζητώ να λάβετε το λόγο και να παρουσιάσετε τα στοιχεία που έχετε να παρουσιάσετε παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρα, κύριε Σβόμποντα, αξιότυπα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα καταρχάς να απευθύνω στον καθένα από εσά έναν εγκάρδιο χαιρετισμό και μία και πραγματικές ε, ευχές ε, για, την, ε, για τις εργασίες της Επιτροπής σας που συστάθηκε πρόσφατα μέσα στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σημαντικής νομοθετικής θητείας για την Ευρώπη. Μια θητεία που κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να επενεξετάσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές όσον αφορά τα συμφέροντα και τις προσδοκίες των πολιτών μας. Η Ιταλική Προεδρία έχει ξεκινήσει το δρόμο της ε, και εργάζεται εν ώψη των επόμενων θεσμικών ε, συναντήσεων. Ε, το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου και η Τρίλογη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας εγγυηθώ την προσωπική μου δέσμευση να αναπτύξουμε μία καρποφόρα συνεργασία ε, στο, ανάμεσα στο Συμβούλιο Τζάι και την Επιτροπή σας για τα θέματα αρμοδιότητας ε, τα, τους επόμενους μήνες. Ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε το ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης ε, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και να λάβουμε υπόψη μας ε, την, ε, τις διαφορές ανάμεσα στις ένομες τάξεις και τις δικαστικές παραδόσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας μέσα στα πλαίσια ε, του προγράμματος το οποίο έχουμε εκπονήσει με τις δύο προεδρίες της Λετωνίας και του Λουξεμβούργου που θα μας διαδεχθούν τους επόμενους 12 μήνες στο Συμβούλιο και που συμμερίζονται απόλυτα τους στόχους μας. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26-27 Ιουνίου τονίζουν ε, όπως όλες οι ε, διαστάσεις μιας Ευρώπης που προσφέρει ουσιαστικά δικαιώματα στους πολίτες της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ε, Ένωσης. Η Ιταλική Προεδρία γνωρίζει απόλυτα ότι η επιτυχία ή η αποτυχία σε έναν τομέα εξαρτάται από την πρόοδο και από τις οπισθοδρομήσεις σε άλλους τομείς και όχι μόνο από τις συνεργίες ε, με τους τομείς ε, τους, που σχετίζονται. Ε, ιδιαίτερα είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι μια στενή συνεργασία ανάμεσα σε μια ε, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα αστικής δικαιοσύνης και ε, και την οικονομική ανάπτυξη. Μόνο η βεβαιότητα όσον αφορά τους κανόνες και η, ευκολία στην πρόσβαση για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις ε, στα διάφορα εργαλεία ε, προστασίας των δικαιωμάτων μπορεί να συνεισφέρει στην υπέρβαση των της δυσπιστίας και των προκαταλήψεων που πολλές φορές αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια ε, στην, ε, στις εξελίξεις και στις επενδύσεις στο ευρωπαϊκό χώρο. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας, το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω, ε, είναι ε, ευθυγραμμισμένο με τις ε, πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο, οδηγίες, δύο οδηγίες με βάση τις οποίες θα οργανώσουμε τις το, το εξάμεινο της Προεδρίας μας είναι η συνεργασία από τη μία πλευρά ανάμεσα στην αστική δικαιοσύνη και στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα και από την άλλη ανάμεσα στην αστική δικαιοσύνη και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι καταρχάς να, διευκολ... να ε, ε, προχωρήσουμε τα θέματα όσον αφορά την ρύθμιση των μικροδιαφορών και την διαδικασία της αφαιρεγγιότητας. Επίσης θέλουμε να εξετάσουμε και τα θέματα που αφορούν τις προτάσεις του κανονισμού για τις ε, συνέπειες στην περιουσιακή κατάσταση όπως ε, διαμορφώνεται μετά από το διάλυση του γάμου ανάμεσα σε διασωνιαριακά ζευγάρια και από την λύση μιας ε, ε, ε, ε σχέσης συμβίωσης. Η πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού 861 το 2007 δημιούργησε μια ευρωπαϊκή διαδικασία για τις, ε, διαφορές, ε, για τις μικροδιαφορές. Πέραν όμως ε, των εργασιών που όσον αφορά την ρύθμιση αυτού του εργαλείου πρέπει να, να προωθήσουμε το εργαλείο αυτό ακόμα περισσότερο. Ε, η διεύρυνση του τομέα της εφαρμογής, ε, η τεχνολογική εφαρμογή των μέσων όσον αφορά την ε, συλλογή των αποδείξεων και την κοινοποίηση των εγγράφων και μια μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αναφορά την κατανομή των δικαστικών δαπανών θα καταστήσει το εργαλείο αυτό για, τις, την επίλυση των μικροδιαφορών δηλαδή πιο ελκυστικό για τους για την πρόταση, ε, ε, με πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, ε, έχουμε δεσμευθεί να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει στη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης τον επόμενο Δεκέμβριο. Όσον αφορά τώρα την πρόταση κανονισμού για την διαδικασία αφαιρεγκαιότητας, ε, ξεκινάμε με την εντολή που δόθηκε ε, από το Συμβούλιο το προηγούμενο εξάμεινο και να θέλουμε να διαπραγματευτούμε με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ε, διαβεβαιώσω την Επιτροπή σας, την Νομική Επιτροπή, ότι η Ιταλία θέλει να υπάρξει μια ουσιαστική πρόοδο στο θέμα αυτό και θα δεσμευθούμε να το, να το εξετάσουμε ε, περαιτέρω. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα, πετύχουμε μια κάποια συμφωνία. Συνειδητοποιούμε ότι το κείμενο ε, του Συμβουλίου περιέχει πολλές, πολλά, πολλές ευαίσθητες ε, αναφορές, κυρίως όσον αφορά την διαδικασία συντονισμού της αφαιρεγγιότητας για τους ομίλους των εταιριών. Ε, επίσης ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την προστασία των εταιριών και των τοπικών πιστωτών ε, που θα πρέπει να που πρέπει να γίνουν σε τέτοιο, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο έτσι ώστε να μην αποτελεί πυρήνα των προσπαθειών μας η χρεοκοπία ενός ε, ε, επιχειρηματία, αλλά αντίθετα η ε, η σωτηρία του και η ανάκαμψη, ουσιαστική ανάπτυξη, ανάκαμψη στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά ε, την πρόταση του κανονισμού σχετικά με την αποδοχή συγκεκριμένων ε, δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης ε, και την κατάργηση της επικύρωσης κάποιων εγγράφων. Η Ιταλική Προεδρία θεωρεί προτεραιότητα την, ε, τις διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα γιατί θεωρεί ότι είναι ένα, ε, μια, σημαντικό στάδιο για να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και την εγκατάσταση των πολιτών και των επιχειρήσεων περιορίζοντας ε, το κόστος η συζήτηση ε, αυτού του θέματος στο άτυπο Συμβούλιο του Μιλάνου της 9ης Ιουλίου με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά του Προέδρου Σβόμποντα και η μεταγενέστερη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο έδειξε ότι υπάρχει μια σαφής θέση από πλευρά των κρατών μελών όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ε, η Ιταλική Προεδρία θέλει, έχει σαν στόχο να επωφεληθεί από την συζήτηση που έλαβε χώρα στο Μιλάνο για να προχωρήσει ταχύτατα τις εργασίες λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ε, χρειάζονται συγκεκριμένους κανόνες και απαιτούν ε, να απελευθερωθούν από τα δεσμά της γραφειοκρατίας που πάρα πολύ συχνά συχνά ε, ε, εμποδίζει να διακινηθούν ε, ελεύθερα από μία χώρα σε μια άλλη και καθιστά την σχέση με τις δημόσιες αρχές ιδιαίτερα προβληματικές. Έχουμε έχουμε καταγράψει μια κάποια ευελιξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των αντιπροσωπιών όσον αφορά το εύρος του πεδίου εφαρμογής. Ε, θα, θα έχω και μία συνάντηση σήμερα με τον Επίτροπο τον κύριο Ράιχετς για να ε, προωθήσουμε τη συνεργασία μας και εν ώψη των ε, επόμενων πρωτοβουλειών που θα αναλάβουμε. Γνωρίζω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπέρ πέρα μιας ε, εφαρμογή ε, του κανονισμού και ελπίζω ότι θα έχω και θετικά μηνύματα ε, και όσον αφορά την μεθοδολογία και όσον αφορά την ουσία της μιας σταδιακής προσέγγισης. Τώρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι ο δρόμος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι δύσκολος και αναφέρομαι στις ανησυχίες κάποιων κρατών μελών σχετικά με το επίπεδο αξιοπιστίας των εγγράφων και των δηλώσεων που προέρχονται από άλλες χώρες. Αλλά ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το λόγο ε, θέλαμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας ε, όσον αφορά τουλάχιστον ένα πρώτο πυρήνα των εγγράφων και αυτό θα αποτελέσει την σπίθα που θα αναπτύξει ε, το μεγάλο δυναμικό το οποίο εμπερικλείεται σε αυτό το εργαλείο συνεργασίας και θα ε, δώσει ένα κίνητρο στα κράτη-μέλη για να ε, συμπεριλάβουν στο μέλλον και ένα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εγγράφων. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουν οι εργασίες τον πιο γρήγορα και για να πετύχουμε με ένα γενικότερο προσανατολισμό μέσα στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Για να ολοκληρώσουμε ε, τον πρώτο κύκλο των εργαλείων αστικής δικαιοσύνης τον οποίο ε, με τον οποίο εργαζόμεθα, ε, θα ήθελα να ε, αναφερθώ και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις πωλήσει. Ε, για τον σχετικό κανονισμό. Ε, παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ψηφοφορία του, της 26ης Φεβρουαρίου που έδωσε ένα σαφές μήνυμα για την ε, επανεκκίνηση αυτού του, του θέματος μέσω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως. Και περιμένουμε τώρα τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως την εξέταση του, ε, του παραρτήματος της πρότασης σύμφωνα με τα συμπεράσματα τα οποία κατέληξε το ε, Συμβούλιο Τζάι τον Ιούνιο του 2012 ε, και θα ήθελα να κλείσω εδώ την, ε, την παρουσίαση του προγράμματός μας ε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ενδυναμώσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών κυρίως στα θέματα που αφορούν το αστικό, την, την αστική δικαιοσύνη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, μια βεβαιότητα, ε, την σαφήνεια του, και την ασφάλεια του δικαίου, να χορηγήσουμε μια εύκολη ή ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην δικαιοσύνη σε περιπτώσεις ε, διασωνοριακές. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, κυρίως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε στο μέλλον, είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων μέσω της κατάργησης των εμποδίων, κυρίως για τους πολίτες που ε, ζουν και κινούνται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι σε δύο προτάσεις ε, που αφορούν τις ε, συνέπειες στην περιουσιακή κατάσταση μετά από την λύση του γάμου και των σχέσεων καταχωρημένης συμβίωσης θα πρέπει βέβαια να λύσουμε και κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη συμφωνία αλλά θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό θα θέλαμε να υποβάλουμε στα κράτη-μέλη νέα σημεία προσκέψη και προσπαθώντας να βρούμε μια κοινή απάντηση που θα επιτρέψει στις προεδρίες που θα μας απασχολήσουν να ε, επωφεληθούν από την δουλειά που έχουμε κάνει. Ελπίζουμε ότι όλοι θα καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ε, νομική ασφάλεια στα άτομα τα οποία, τα, ε, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές χώρες και τα οποία παντρεύονται, γιατί θέλουμε ακριβώς να εξασφαλίσουμε καλύτερα την προστασία των πολιτών. Επίσης, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Ε, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και στο, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη ε, έχουμε συζητήσει κάποια θέματα τα οποία ξέρουμε ότι θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα τις εργασίες εφαρμογής της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης ε, πάνω στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία γνωρίζει απόλυτα τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε για να πετύχουμε έναν ουσιαστικό χώρο, ε, ουσιαστικό ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, ένα χώρο ελευθερίας και ασφάλειας, όπου οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα τα δικαιώματά τους σε κάθε γωνιά της ευρωπαϊκής επικράτειας. Είμαστε Γι' αυτό ε, υπέρ μιας ε, στενής και ουσιαστικής και ειλικρινούς συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχει τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας όσον αφορά τις προτεραιότητες τελικής προεδρίας καθώς επίσης σε θέματα που έπρεπε της αρμοδιότητας της Δημιάς Επιτροπής. Εάν μας επιτρέπετε τώρα κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος αυτά τα οποία είπατε μόλις εκφράσατε συνάδουν με την απόψεις πλειοψηφίας αυτής της Επιτροπής όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δικό μας τομέα και τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη αυτής της Επιτροπής για να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων αυτών. Πρώτος είναι ο κύριο Καβαντά είναι ο πρώτο στην κατάλογο των ομιλητών, των αγορητών. Παρακαλώ κύριε Καβαντά για το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. κύριε Υπουργέ, Έρχεσαι στην Προεδρία σε ένα κόντεξ το οποίο πραγματικά δεν είναι κανονικό, δεν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα κανονικό αλλά είναι έκτακτο και το οποίο πραγματικά πρόκειται περί διακοπής της ιστορίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη εστράφει εναντίον και αντιτίθεται στην ειρήνη και στην ευμερία της Υπήρου μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά περί τίνος ομιλώ και γνωρίζετε ότι και στη χώρα σας ακόμη έχουν πάρει ε, ένα μέρος των ψήφων ακόμη και στην Ιταλία και δεν απόκειται σε μένα ε, σαν Γάλλο, όχι σαν Γάλλο μόνο αλλά σαν Ευρωπαίο Γάλλο που θα σας δώσω ένα μάθημα διότι εμείς στείλαμε το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που προσμένο από την Ιταλική Προεδρία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο στο πνεύμα μου, στο σώμα μου και στην καρδιά μου είναι πολύ ευτυχή συγκυρία διότι η χώρα σας βρίσκεται σε μία, σε μία νέα παλιγενεσία θα έλεγα ξέρετε ότι πέθανε η χώρα σας πάρα πολύ στην εσωτερική πολιτική όσον αφορά τον έξι ξεχρονισμό του κομμουνισμού, ε, όλον εκείνο το λαϊκισμό τον οποίο κληρονομήσατε μέχρι τώρα. Η προεδρία σας λοιπόν είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη χώρα σας αλλά και στην Ευρώπη παρά το γεγονός ότι προσμένουν τέσσερις μήνες ωστόσο προσμένουμε πάρα πολλά και έκτακτα πράγματα και εκπληκτικά πράγματα εκ μέρους σας. Τα σημεία τα οποία υπογραμμίσατε ε, ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικά και όταν ακούω τον κύριο Ρέντζη τον πρωθυπουργό σας του οποίου ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας εξέπληξε όλους ευτυχώς θα ήθελα να σας ζητήσω χωρίς να αμφιβάλλω όσον αφορά τις προτεραιότητες σας παρακαλώ να καλύψετε όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν ναι. Και να βάλετε όλη τη δύναμη σας σε αυτό και ιδιαίτερα σε δύο τομείς. Πρώτον, να προσπάθ, να βάλετε σε μια τάξη και σύμφωνα με τις γενικές αρχές αλλά και το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή την επιτρομή ε, η δική μας επιτροπή είναι η αρμόδια επιτροπή χώρες εκείνες οι οποίες πραγματικά δεν ακολουθούσαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε, έκαναν κατά το δοκούν και ιδιαίτερα σε χώρες εκείνες που βρίσκονται στο, κοντά στο Δούναβι όσον αφορά την οργάνωση και την οργάνωση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει να υπέρθει τάξη σε αυτό τον τομέα. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το τονίσετε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να σας υποβάλω, σας συμβολή πρόεδρα μου και μου, ε, κύριε Υπουργέ, και δεν είμαι ο μόνος κύριε πρόεδρε, δεν είμαι, είμαι ο πρώτος ο μιλών, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Θα ήθελα η δράση σας λοιπόν και χάρη στη νιώτη σας και χάρη σε όλο το ιστορικό σας και την κυβέρνηση στην οποία ανήκετε θα πρέπει να δράσει άπαξε διαπαντός ενάντια της εγκληματικότητας με καλύτερη δυνατότητα ανακρίσεων, παρακολουθήσεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν για διαπραγματεύσει όσον αφορά την ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα λέγω όχι γιατί θέλω να σα κάνω μάθημα, κύριε Υπουργέ. Και γνωρίζετε κάλλιον μου την ε, δυσκολία αλλά και το επικίνδυνο του χαρακτήρου αυτής της εγκληματικότητας και πόσο μάλλον που η χώρα σας είναι μεταξύ των θυμάτων αυτής της εγκληματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίζουμε στη δική σας ε, Προεδρία και σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός σας για το θέμα αυτό ούτως ώστε να εξαφανιστεί οποιαδήποτε ανομαλία η οποία υπάρχει στον τομέα της εγκληματικότητας, τα οποία, η οποία εγκληματικότητα αυτή τη στιγμή έχει δράσει πάρα πολύ αρνητικά όσον αφορά την Ευρώπη και την οπτική που έχουν οι άνθρωποι για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Καβαντά. Επόμενος, ο κύριος Ζιεύκοφ. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο τον οποίο εκφωνήσατε, ο οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και έχει ε, ουσία και περιεχόμενο. Ήταν κάτι που ανέμενα εγώ. Τα θέματα τα οποία επιλέξατε και τα οποία παραθέσατε, απαριθμίσατε και επί των οποίων εργαζόμαστε είναι θέματα τα οποία είναι μέσα στα, ήταν στην ε, ημερήσια διάταξή μας αλλά παραμένουν και κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Η Επιτροπή μας είναι αλλού διαφορετική από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι μια επιτροπή η οποία όντως επιστιάζεται σε, στο περιεχόμενο κάνει μια εργασία η οποία είναι θετική για την ανάπτυξη δικαιωμάτων των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει. Δημιουργώντας λοιπόν ζώνες ασφαλείας στην Ευρώπη και αυτό πραγματικά. Όσον αφορά τις ελευθερίες βέβαια είναι και η Επιτροπή των ε, Ανθρωπίνων Ελευθεριών. Και βέβαια σε αυτό το σημείο μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μόνο και ημών. Επίσης υπογραμμίσατε πόσο σημαντικό είναι να, να περατώσουμε όλα αυτά, όλους αυτούς τους φακέλους, τα δοσία τα οποία έχουμε, τα οποία, τα οποία θα πρέπει να λυθούν διότι έχουν επιπτώσει επί των οφθαλμών των πολιτών μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αφηρημένοι, αφηρημένοι νόμοι. Σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε τους πολίτες μας και να υπάρξει μια ειρηνική διευθέτηση των θεμάτων αυτών, θεμάτων, τα θέματα της κοινή ιδιοκτησία σε γάμους είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό την κατανομή του στη διάθεση αυτών των ε, θεμάτων και την επίλυση του, καθώς επίσης τη δυνατότητα να υπάρχουν όλα τα κείμενα μεταφρασμένα και αναγνωρισμένα επαρκώς. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας όταν λέτε ότι η όλη διαδικασία να υπάρχουν ε, έγκυρα κείμενα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε το επιφυκτό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο αυτός ο στόχος είναι μεγάλος ή τεράστιος ή ευρύς αλλά ωστόσο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες και όπου τα, όλα τα κρατη θα μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, και θα πρέπει να περιλαμβάνουμε και περισσότερα έγγραφα σε αυτόν τον κατάλογο. Για να ανακεφαλαίωσω λοιπόν με τις προτεραιότητες τις οποίες αναφέρατε θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις εργασίες όσον αφορά τη δίκαιο τους πτώχευσης, το θέμα της φερενκιότητος και θα έχω τη χαρά να είμαι εισηγητή σε αυτά τα ιδιαίτερα ντοσιέ θέματα και το ερώτημά μου θα είναι το εξής κύριε Υπουργέ πόσο πραγματικά θα πρέπει να βρούμε χρονοδιαγράμματα ε, προθεσμίες όπου πραγματικά μπορούν να επιτελεστούν αυτά τα πράγματα με τις ανακατάλληλες συζητήσεις και τροπολογίες οι οποίες θα γίνουν και πιστεύω να περατώσουμε αυτές τις εργασίες κατά τη διάρκεια της Ιταλικής, Ιταλικής Προεδρίας. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές απόψε αυτό το θέματος και μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και θα σας στήσω να διασφαλίσω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το μέγιστο για να κλείσουμε αυτό το φάκελο ώστε όλοι να είμαστε ευτυχείς εν τελική αναλύση. Αύριο θα ξεκινήσουμε σε αυτό το θέμα και πιστεύω πως ο κύριος δεν είναι ένας από τους ηγητές μας και ο κύριος Μπελίνγκουερ και προφανώς μερικοί νέοι συνάδελφοι οι οποίοι αναλαμβάνουν με τη σειρά τους αυτό το φάκελο. Νομίζω κάναμε μεγάλο δρόμο, μακρύ δρόμο σε αυτό το θέμα και είναι καιρός να το περατώσουμε. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο δεν είναι τόσο αποφασισμένο για αυτό το θέμα. Άρα βρίσκεται η μπάλα στο δικό σας γήπεδο και ευελπιστούμε πως θα περατωθεί η υπόθεση, θα παίξουμε το παιχνίδι, λέει ο Σαν υπουργό ε, δικαιοσύνη, το Υπουργείο Δικαιοσύνη είναι ένα βασικό Υπουργείο κλειδί, θα έλεγα. Αυτό είναι ο για τον οποίο ότι η τελική αναλύση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα νομοθέτημα δεδομένο, συγκεκριμένο και μερικέ φορέ ενώ αυτά γίνονται μερικά κράτη, δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτή τη νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια καμπάνια, μια εκστρατεία για πληροφόρηση εκ μέρου τη Κομισιόν και αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί και από την επόμενη Προεδρία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε αυτή η πληροφόρηση να φτάσει στου πολίτε μα και είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω πως αυτό θα είναι ένα μέσο διευκόλυνση της καταστάσεω, όχι μόνο για, τον, για το κράτος αλλά καθώ επίσης τι λύσει δώσαμε, πώς επιλύσαμε τα προβλήματα στα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτε μα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν νέες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προτεραιότητά σας και υποστηρίζω πλήρως αυτές που σε εκφράσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος αγορητής, κυρία Ράγκνερ. Κυρία Ράγκνερ λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζουμε τερμά και ευχαριστούμε πολύ που παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας, κύριε Υπουργέ. Η Ιταλική Προεδρία ε, συμπίπτει με, μια ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή ε, εξελέγησαν οι ευρωβουλευτές, ε, θα έχουμε σύντομα μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντωμεταξύ θα έχουμε και την τελική Προεδρία η οποία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τη συνέχεια. Θέλω λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου στα εξή θέματα. Καταρχήν πολύ σύντομα όσον αφορά τα πιστοποιημένα έγγραφα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη κατά την προηγούμενη θητεία ασχολήθηκε, ε, επιλήφθηκε του θέματος, ε, προσπάθησε να βρει μια λύση φιλική προς τον πολίτη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστούν για αυτό το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει ε, πιο συγκεκριμένα τι θα γίνει τελικά με τα πιστοποιημένα έγγραφα. Το δεύτερο που θέλω να πω, η Ιταλική κυβέρνηση και τώρα αναφέρομαι στην κυρία Μογκερίνη. Η Ιταλική κυβέρνηση έδειξε λοιπόν με την επιλογή της κυρίας Μογκερίνη ότι επιθυμεί ε, διακαώς να προάγει ε, της, ε, τη θέση των γυναικών. Αυτό συνδέεται άμεσα και με τη θέση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Νομίζω η Ιταλική Προεδρία κατέδειξε σαφή στάση στην δική μας την Ολομέλεια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Η Ιταλική Προεδρία, αυτό το θέμα το οποίο όπως σας είπα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ολομέλεια, πώς προτίθεται να το προάγει. Γιατί βεβαίως αυτό το θέμα έχει άμεση σχέση και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λευκατόν. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την έκθεση ενδιαφέρουσα και πολύ ευγενή. Λυπάμαι που ο κύριος Καβαντά είπε πράγματα που δεν υπήρξαν ε, ευγενικά αλλά υβριστικά θα έλεγα ε, εναντίον ορισμένων βουλευτών ένιωσα να στοχεύομαι με αυτά τα οποία είπε γιατί εγώ είμαι πατριώτης κύριε Πρόεδρε τι κατάλαβε να μου πει ο συνάδελφός μου για να μου πει ότι τον εξέβρισα αλλά δεν πειράζει σας αντιλήφθη κύριε Καβαδά χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς ε, κι άλλα λόγια ευριστικά κύριε Καβαντά μου λέτε έτσι λοιπόν θα ήθελα να θέσω σαφείς ερωτήσεις στον κύριο Υπουργό όσον αφορά ένα μέρος της παρουσίασής του. Υπογράμμισε ότι θα ήθελε να ευνοήσει έναν κανονισμό μικρών διαφορών που δημιουργούνται. Είναι ένα θέμα το οποίο με διέφερε τα μάλα στην παρουσίασή του και φρονώ αυτός ο κατάλογος εργασίας μπορεί να είναι κάτι καλό βεβαίω καταρχήν, αν υπάρξουν προτώσεις οι οποίες όπως ανέφερα θα υπάρξουν και ωστόσο υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ενάντια της, της σπουδής της ε, δικαιοσύνης. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που έχουν σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, δια μια δικαιοσύνη η οποία δύο τα μια ταχύτητα η οποία πηγαίνει αργά για τα κοινά θέματα και άλλα που πάει υψηλή ταχύτητα εφόσον υπάρχουν εμπλεκόμενα συμφέροντα. Υπογραμμίζω λοιπόν τον κίνδυνο που υπάρχει σε αυτή την προσέγγιση. Δύο ερωτήσει λοιπόν που θέσω. Όταν εσείς αναφερθήκατε προηγουμένω σε μικρές διαφορές, τι εννοείτε με λέξεις μικρές διαφορές. ποια είναι η μικρή διαφορά και η δεύτερη ερώτηση, τι καλείται επιτάχυνση, αυτή η διαδικασία επιτάχυνσης. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι θα πάει πολύ πιο γρήγορα διαδικασία στα κανονικά δικαστήρια ή εννοείται ότι θα αναλάβετε ορισμένε αρμοδιότητε αρμοδιότητες από τα τακτικά δικαστήρια τα σημερινά. Ευχαριστώ. Τέλος. Ο κύριος Δαδιαφιωμή είναι ο τελευταίος αγορητής στον καταλογό μου. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που παρουσιάσατε στον Ιούνιο είναι σημαντικά. Ξέρετε, από την αρχή της χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε παιδιά υιοθέτησε μερικά πράγματα όσον αφορά τους, την κοινή νομοθεσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εμπόρους καθώς επίσης και από τους καταναλωτές και το οποίο αντιτίθεται οποίες διαφορετικά από 28 ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτό ή οι καταναλωτές, παρόλα αυτά η πρόταση αντιμετωπίζει αντίσταση από ορισμένε κράτη στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Υπάρχει λοιπόν αντίσταση όσον αφορά των διοικητικών αυτών μέτρων, πράγμα το οποίο είναι κατά των συμφερόντων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να απαντήσει τα ερωτήματα τα οποία έδωσα. Κοιτάξτε, Όσον αφορά στο θέμα το οποίο έθιξε ο Αντιπρόεδρος κύριος Καβαντά, θα ήθελα να πω ότι ε, να είστε σίγουροι ότι για μας είναι πολύ σημαντικά τα θέματα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ιταλία πιστεύει ότι αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Η Ιταλική Προεδρία έχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλους εκείνους ε, τους ε, πολιτισμούς που ε, υπήρξαν ιδρυτικά στοιχεία της σύμβασης, της ιδρυτικής σύμβασης. Αυτά όσον αφορά και τα τις αρχές που πρέπει να ισχύουν στα κράτη-μέλη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διαβεβαιώσω τον κύριο Αντιπρόεδρο για την πρόθεσή μας με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό ένταλμα δηλαδή να προκύψει ένας ε, οργανισμός ε, που να είναι ανεξάρτητος παρότι πρέπει να σας πω ότι εδώ προσκρούμε σε πολλές αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη θεωρώ όμως ότι κάτι τέτοιο είναι καθοριστική σημασίας για να υπάρχει πραγματικά ουσιαστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και θα ήθελα να σας πω και το εξής, ότι και η δουλειά αυτής της Επιτροπής είναι καθοριστική σημασίας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οι, τα κράτη-μέλη, οι σχετικές νομοθεσίες ε, βασίζονται στο ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που έχει προκύψει και ο ρόλος που διαδραματίζει το οργανωμένο έγκλημα. Οι ιδιοκτικέ αρχές είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως εγώ πιστεύω ότι η αστική δικαιοσύνη δυστυχώς ε, έχει υποτιμηθεί σε σχέση με την αντιμετώπιση ε, του προβλήματος του οργανωμένου εγκλήματος. Όσον αφορά τώρα στο θέμα της ε, νομιμοποίησης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς προτιθέμεθα να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Επιθυμούμε να ε, συμφιλιώσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτή του Συμβουλίου. Και ας ξεκινήσουμε με τα θέματα όπου υπάρχει συμφωνία. Εδώ λοιπόν επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην εισήγησή μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασίας από κοινού να κάνουμε το πρώτο βήμα να δούμε πού ακριβώς έχουν οριμάσει τα πράγματα για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και πιστεύω ότι είναι και καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καθορίσει ένα χάρτη πορείας ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στην ε, εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Πάντως ε, σήμερα υπάρχει κινδύνος ε, να καταλήξουμε σε αυτό που λέμε ε, το τέλειο είναι ο εχθρός ε, του καλού. Δηλαδή να θέλουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε στα κράτη-μέλη. Και είναι δύσκολο να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί όταν θα υπάρξει το πρώτο έγγραφο το οποίο θα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλα τα κράτη-μέλη, τότε νομίζω ότι αυτό θα τύχει της ε, θετικής αντιμετώπισης από την κοινή γνώμη και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και τότε αυτό θα μπορούν να το ε, αντιμετωπίσουν ως ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει τη ζωή τους και τις οικονομικές ε, συναλλαγές όπως έγινε δηλαδή και με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς το σημαντικότερο είναι να γίνει το πρώτο βήμα και μετά να ακολουθήσει μια σταδιακή πρόοδος. Κατόπιν, ας πάμε τώρα στο θέμα της ισότητας ε, των δύο φύλων. Ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν εμπίπτει στις δικές μου τις αρμοδιότητες. Είναι όμως σαφές ότι η Ιταλία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό ξεκινάμε αν θέλετε και από την κυβέρνησή μας, από το πώς έχει επανδρωθεί από την ε, συνεισφορά και των ανδρών αλλά και των γυναικών ε, στην, ε, στα διάφορα καθήκοντα στα δικά μας τα Υπουργεία και στα αξιώματα της κυβέρνησής μας προάγονται πρωτοβουλίες κοινωνικής φύσεως στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών ακριβώς για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης και βίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό ε, να επισημάνουμε το πόσο σημαντικά σας είπα είναι όλα αυτά τα θέματα για τη δική μας την κυβέρνηση. Μας ενδιαφέρει να, υπάρχει, να υπάρχουν πιο κατάλληλα εργαλεία κυρίως όσον αφορά ε, περιπτώσεις βίας εις βάρος των ε, γυναικών. Όσον αφορά τώρα στα περίφημα small claims, στις μικρές διαφορές. Θέλουμε να βρούμε κάποια λύση. Και θέλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος της ε, χρήσης δύο ταχυτήτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι, εν πάση να υπάρξει κάποια μετακίνηση. γιατί το να θέλει κανείς ε, να προστατεύσει κάποια δικαιώματα πολλές φορές αυτό και μόνο ενέχει κάποιες αντιφάσεις σε όλα τα κράτη, ε, μάλλον υπάρχουν διαφορές ε, ανάλογα με τα, με τα κράτη-μέλη. Ε, θεωρώ όμως ότι δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε αυτή τη συζήτηση και αυτό θα το προσέξουμε ιδιαίτερα όσον αφορά, σας είπα, το σύστημα της παροχής εγγύσεων. Για το θέμα των φορέων αυτό είναι ένα από τα θέματα όπου τα κράτη-μέλη έχουν κάποια δυσκολία ε, να επιτύχουν μια μορφή ισορροπίας. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία εξετάζουμε. Είναι θέμα Συμβουλίου το να κατατεθεί μια σχετική σύσταση. αναφέρομαι στο θέμα των φορέων κάτω από το πρίσμα των μικρών διαφορών. Δηλαδή ε, ότι θα πρέπει κανείς ε, να έχει κατά νου ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα τα οποία κατά κάποιο τρόπο παρακάμπτουν τη νομοθεσία. Ακόμα και αν υπήρξαν κάποιες εξοδικαστικές μορφές αντιμετώπισης των προβλημάτων και των διαφορών. Νομίζω ότι πάντα υπήρχε δυνατότητα της δικαιοσύνης ε, να παρέμβει. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος να αποκλίνει από αυτά, αυτές τις βασικές αρχές. Θεωρώ ότι πρόκειται εδώ για θεμελιώδεις αρχές ε, του κράτους δικαίου για προπύργια, αν θέλετε πιο χαρακτηριστικά, του κράτους δικαίου. Κατόπιν, όσον αφορά στο θέμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου περί πολίσεων, ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερα στη δική μου την έκθεση και να διευκρινίσω τα στοιχεία αυτά. Το Συμβούλιο λοιπόν εξετάζει το παράρτημα της πρότασης και της εργασίας του της ε, βασίζει στις, ε, ε, Συμβουλίου Γκάιντελ του 2012 του Συμβουλίου Τζάι περί εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρώσουμε όπως ε, σας είπα ε, τις προτάσεις κατά τη διάρκεια της Ιταλικής ε, Προεδρίας. Εμείς παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτού του θέματος και στην Ολομέλεια της 26ης Φεβρουαρίου είδαμε ότι εκεί προτείνεται διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εξ αποστάσεως ε, πωλήσεων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει πάρα πολλές ε, δυνατότητες ε, για την ενίσχυση της κοινή αγοράς. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά εκ μέρους όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Και εμένα πρέπει να σας πω, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι Υπάρχει κοινή αντιμετώπιση κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Ε, θα συνεργαστούμε για να αναζητήσουμε μια συμφωνία γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο τομέας ε, είναι καθοριστικής ε, σημασίας. Άρα δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία κυρίως για τις πρωτοβάθμιες υποθέσεις που εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι, σε, ότι αυτές οι εξελίξεις είναι καθοριστικής σημασίας έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη ισχύ της δικαιοσύνης. Αλλά ε, και να μπορούμε επίσης να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε κάποια δικαιώματα. Κατόπιν τούτου η δική μας η δουλειά είναι ότι θέλουμε να ακούσουμε καταρχήν τις απόψεις όλων εκείνων που ασχολούνται με το θέμα για όλα αυτά τα χρόνια και να ακούσουμε και την άποψη της αρμόδιας επιτροπής. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια συνάντηση στην ε, Ρώμη που όπως σας είπα η συνάντηση αυτή θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλετε, όπως επίσης ε, και για όλα αυτά τα οποία είπατε σχετικά με το ρόλο ε, και τις αρμοδιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Από όλα αυτά που ακούστηκαν ε, καταλήγω στο ότι έχετε πάρα πολλές ε, προσδοκίες και ελπίζουμε εμείς να μην σας απογοητεύσουμε. Πάντως η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ρεαλισμός με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εξετάσει τα θέματα που έχουν τεθεί, η αποφασιστικότητα θα είναι καθοριστική και η συνεισφορά του Κοινοβουλίου θα είναι καθοριστική σημασία για να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι που έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια τη δική μα Προεδρία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της Ιταλικής Προεδρίας ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε ότι ήταν και πολύ καρποφόρα ε, ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας. Ladies and we Μετά τον Υπουργό κύριο Ορλάντο έχουμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Υφυπουργό ε, της Ιταλικής Κυβέρνησης ε, για τα ευρωπαϊκά θέματα, τον κύριο Σάντρο Γκότσι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να, μας και να σας ζητήσω να μας πείτε ε, κάποιες από τις προτεραιότητες της τελικής ε, Προεδρίας που αφορούν την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ε, είμαι πολύ χαρούμενος που σας συναντώ, που σας γνωρίζω σε αυτή την αρχή της ε, θητείας. Ε, η Ιταλική Προεδρία θέλει να ξεκινήσει ένα νέο πολιτικό κύκλο που θα επικεντρωθεί σε λιγότερες προτεραιότητες αλλά πολύ περισσότερο σημαντικές. Γιατί για μας ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα νομικά θέματα, για τα νομοθετικά θέματα που αποτελούν ε, και τον πυρήνα των εργασιών της Επιτροπής σας κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και όλα αυτά ε, από την σκοπιά της ε, απλούστευσης. Θέλουμε ακριβώς να ολοκληρώσουμε το έργο, να το συμπληρώσουμε, να το απλουστεύσουμε και γύρω από αυτά ε, τα θέματα γυρνάνε όλες μας οι πρωτοβουλίες και οι προτεραιότητες. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Ιταλικής ε, Προεδρίας θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, στενά κυρίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την προστασία των δικαιωμάτων και, την, και, να, ε, και να ευνοήσουμε τις διασυνοριακές ε, ε, συναλλαγές. Αυτά είναι τα τρία θέματα, οι τρεις τομείς τους οποίους θέλουμε να προωθήσουμε και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε στενά για να προχωρήσουμε. Και επίσης Υπάρχει η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του know-how, η ελευθερία της ε, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη νομοθετική εργασία που πρέπει να γίνει και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να προετοιμάσουμε τις συνθήκες ε, για να έχουμε μια πραγματική πολιτική η οποία θα είναι στραμμένη προς την ανάκαμψη και, να, και στραμμένη στην ε, στην ανάγκη να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις ε, στους ε, πολίτες, διότι όντως πρέπει να δώσουμε μια νέα πνοή. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα θέματα και όσον αφορά την εσωτερική αγορά αλλά και όσον αφορά την, τα όργανα, τα εργαλεία που χρειάζομαστε για την governance, για τη διακυβέρνηση. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά και το νομοθετικό έργο, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να υιοθετήσουμε νομοθετικά κείμενα τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη και στην βελτίωση του ανταγωνιστικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται να ολοκληρώσουμε και να ενισχύσουμε ε, τα όσα υπάρχουν ήδη κυρίως όσον αφορά τα, το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς, ε, τους κανονισμούς ε, που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι καινούριο θέμα, αλλά είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, έστω και αν στο παρελθόν, ε, στις παρελθούσες θητείες, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά. Διότι και εμείς ε, τώρα ε, δεν το κάνουμε διότι δεν θέλουμε να ε, καινοτομήσουμε, αλλά γιατί ακριβώς πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες, περισσότερες απαντήσεις. Πρέπει να προωθήσουμε την ανάκαμψη, να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και από νομοθετικής πλευράς για να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τους επόμενους εβδομάδες ε, υπάρχει μια σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει σε κάποιους τομείς ε, κλειδιά ε, σε τομεί συνεργασία ανάμεσα στην, στο Συμβούλιο και, στην, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα αναφερθώ σε αυτές, σε αυτές τις πρωτοβουλίες μας. Καταρχάς είναι τα εργαλεία διακυβέρνησης. Προφανώς πρέπει να ε, προωθήσουμε και να βελτιώσουμε την government στα θέματα ανταγωνιστικότητας και εσωτερικής αγοράς. Ε, και ήδη έχουμε κάνει πολλά για να ενδυναμώσουμε τον ρόλο και για να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Κατά την άποψή μας στις δραστηριότητες αυτές υπάρχει και μια διαδικασία ε, που αφορά την αναθεώρηση γιατί χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική και πολιτική για την Ευρώπη του 2020. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο του Μαρτίου του 2015 θα πρέπει να υιοθετήσει μια νέα στρατηγική για το 2020 όμως αυτό απαιτεί να γίνει και μια δουλειά προετοιμασίας, ε, ε, πρέπει να ε, προετοιμαστούμε και μέχρι τότε θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και ελπίζω να τα κάνουμε μαζί για να καταλήξουμε σε αυτή τη νέα στρατηγική του 2020 η οποία θα εστιαστεί στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη τώρα έχει μια άλλη μερίσια διάταξη για να βγει ακριβώς από την ε, κρίση ε, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής, ο jean Κλόντου Γιουνκέρ, έκανε κάποιες δηλώσεις πριν ακόμα ε, επιβεβαιωθεί η θέση του ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την στρατηγική 2020, θα πρέπει να δούμε τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες ε, στρατηγικές αυτές, κατά την άποψή μας, περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο Van Rompuy. Και λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να άρουμε τα εμπόδια τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε νομικό επίπεδο όσον αφορά την εσωτερική αγορά υπάρχουν εμπόδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και 20 χρόνια από τότε που πρωτοανακοινώσαμε την ε, ίδρυση της ε, κοινή αγοράς. Υπάρχουν εμπόδια σε διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένε που θέλουμε να προάγουμε και που δίνουν μια συγκεκριμένη απάντηση όσον ε, αφορά ε, καλύτερο και ευνοϊκότερο πλαίσιο κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διασυνοριακές ανταλλαγές τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο και ε, να αντιμετωπίσουμε κάποιες νέες προκλήσεις. Ε, Υπάρχουν πολλά νομοθετικά και νομικής φύσεως προβλήματα και στην ε, τεχνολογική πρόοδο. Έχω, ας πούμε, κατά νου το θέμα της ε, διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν την διανοητική ιδιοκτησία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είναι ένα θέμα καθαρά νομικό αλλά ε, και νομικό και οικονομικό Ανάλογα βέβαια με τις επιλογές τις οποίες θα κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εξακολουθούν όπως σας είπα να απομένουν πάρα πολλά εμπόδια, φραγμοί στις ε, ανταλλαγές κάτω από το πρίσμα της κοινή αγοράς. Αυτούς τους φραγμούς πρέπει να τους καταργήσουμε και για να γίνει αυτό απαιτείται νομοθετικό έργο. Είναι η δουλειά που ξεκίνησε από την προηγούμενη θητεία και εμεί θεωρούμε ότι κατά διάρκεια αυτής της θητείας πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η εργασία αυτή. Γιατί όπως είπα ότι θα πρέπει να έρθουν τα εμπόδια τα οποία είναι ρυθμιστικής φύσεως, γραφειοκρατικής φύσεως και έχουν σωρευτεί ε, στην εργασία, στο, στη δουλειά και τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου και οι τρεις ε, θεσμοί αναφέρονται στην ανάπτυξη. Θέλουν να έρθουν ε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια κατά τα επόμενα έτη. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. Υπάρχει απομάκρυνση από την Ευρώπη, υπάρχει απογοήτευση και των οικονομικών φορέων. Είχαν πολλές προσδοκίες απέναντι στην κοινή αγορά και δεν ε, εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους ε, αυτές. Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται ότι στην Ευρώπη πολύ συχνά υπάρχουν βραδύτατοι ρυθμοί για την επίτευξη των στόχων. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρξουν διαδικασίες ολοκλήρωσης και απλούστευσης. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο αφορά στο θέμα της governance, ε, της περίφημης διακυβέρνησης και το είπα στην αρχή της παρέμβασής μου. Εμείς πιστεύουμε ότι κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ε, θα υπάρξουν προεκτάσεις από τις δραστηριότητες αυτές. Ελπίζουμε θετικές στις σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έχουμε καταθέσει μία πρόταση ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα στο Μιλάνο την προηγούμενη εβδομάδα. Η πρότασή μας ήταν να βελτιωθεί η governance στον τομέα της ε, ανταγωνιστικότητας, να βελτιωθεί η λειτουργία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που για μας είναι ο πρώτος συνομιλητής κυρίως όταν μιλάμε για νομοθετικές δραστηριότητες. Εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτό το Συμβούλιο υπήρχε πολύ μεγάλη κατάτμιση. Ε, πρέπει λοιπόν ε, αυτή η κατάτμιση και η ασυνέπεια να ε, καταργηθούν Αναφέρομαι πάντα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και στις δραστηριότητες του σχετικού συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τη λήψη αποφάσεων και να διευκολύνουμε και τις ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις για τα πραγματικά προβλήματα κλειδί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και αυτό πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό, σε πολιτικό επίπεδο όπως σας είπα στο Συμβούλιο στις, ε, σε επίπεδο Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και δέσμευση των Υπουργών σε αυτό το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Κατόπιν τούτου ε, να, βελτιωθεί, <coughs> να βελτιωθούν οι εργασίες του Συμβουλίου αυτού που έχουν σχέση με την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, πήραμε λοιπόν εντολή την προηγούμενη εβδομάδα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να βελτιώσουμε την governance ε, τόσο σε επίπεδο τεχνικών ομάδων εργασίας όσο και σε επίπεδο ε, υπουργών, σε υπουργικό επίπεδο εργασίας. Η συμμετοχή και οι σχέσεις με τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, βελτιωθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό συντονισμό. Αυτό αφορά κάποιες συγκεκριμένες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Αντοκονιστικότητας. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν σχέσεις και συναντήσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τελικά να προκύπτουν ε, συζητήσεις ουσιαστικές για μεγάλα θέματα προσανατολισμού, θέματα ανταγωνιστικότητας με τα οποία ασχολούνται και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια σχετική πρόταση την οποία έχουμε συζητήσει, τη συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όπως σας είπα πήραμε την εντολή ε, να καταθέσουμε πιο λειτουργικές ε, προτάσεις και αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι με βάση αυτά που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, το οποίο ζήτησε να ε, διατηρηθεί το πρόγραμμα REFIT και εμείς ε, επιθυμούμε να προωθήσουμε την ε, ρυθμιστική απλούστευση του νομοθετικού έργου. Η δική μας η πρόθεση ως Προεδρία είναι να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της, ε, των ρυθμίσεων και αυτά να γίνουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό είναι έτσι ένα γενικότερο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο και μέσα σε αυτό ε, θα ήθελα να εντάξω συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Και νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές σας ενδιαφέρουν και θα θέλατε να τις συζητήσετε με την Προεδρία. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις ε, προτάσεις είναι αναμφίβολα το θέμα της ε, αναπομπής της ε, οδηγίας ε, που αφορά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και στο εμπορικό σήμα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε πάρα πολλά να επιτύχουμε. Ένα από τα θέματα το οποίο είναι σημαντικό είναι γενικά τα εμπορικά σήματα στην Ευρώπη, το θέμα της ετικετοθεσίας. Και εδώ φτάνουμε και πάλι σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή στην απλούστευση. Επιθυμούμε να είναι πιο εύκολη η προστασία των σημάτων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για να προάγουμε την ανάπτυξη ε, πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα σχετικά με την αναπομπή όλης αυτής της σχετικής ε, νομοθεσίας. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε λιγάκι και τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ε, βλέπουμε εκεί ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, χρησιμοποιούν τα σήματα αυτά την περίοδο 2008-2010 αυτές οι επιχειρήσεις ε, παρουσίασαν το 21% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους αντιστοιχεί δηλαδή το 21% της συνολικής απασχόλησης. Μιλάμε για πάνω από 45 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, περίπου το 34% του ΑΕΠ. Και ε, νομίζω ότι αν υπάρξει συγκεκριμένη συνεισφορά ε, στην εμπορική ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ε, όπου θέλουμε να παρουσιάσουμε νομοθετικό έργο. Βεβαίω έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα διάρκεια της ελληνικής, της λιθουανικής και της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τον Ιούλιο ανέθεσε ή έλαβε την εντολή από το Συμβούλιο ε, να υπάρξει τριμερής ε, συζήτηση για να υποβληθεί συγκεκριμένο κείμενο. Άρα δηλαδή εμεί είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας και ελπίζουμε πριν από την εκπνοή της Προεδρίας μας να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα, μία άλλη σημαντική νομοθετική προτεραιότητα ε, στην οποία θέλω την οποία θέλω να σε επισημάνω είναι η πρόταση ε, οδηγίες που αφορά τα εμπορικά μυστικά. Και σας είπα ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων μας είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε και με θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία διακυβεύονται σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ε, το θέμα της ελευθερίας ε, και διάδοσης θεμάτων ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το, την εμπορική τεχνογνωσία. Υπάρχει η συμφωνία TRIPS που όπως πολύ καλά γνωρίζετε που είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς ως Προεδρία είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες εναρμόνισης γιατί με τον τρόπο αυτό κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσφέρουμε την απαραίτητη προστασία και ε, σε περίπτωση ε, απάτης ή ε, παράνομης χρήσης των ε, εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών θα προστατεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε τις ε, διασυνοριακές ανταλλαγές. Το νομοθετικό έργο θα δώσει όθηση στην έρευνα και την ανάπτυξη, κυρίως ε, στις διασυνοριακές συναλλαγές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Και αυτό θα βοηθήσει τους ε, ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με ε, θέματα έρευνας και ανάπταξης. Αυτά λοιπόν ε, είχα να πω σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Η Ελληνική Προεδρία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τις 26 Μαΐου του 2014 επιτεύχθηκε έτσι ένας ευρύτερος προσανατολισμός επί, επί ενός συμβαστικού κειμένου. Και εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε ε, έγκαιρα το κείμενο και ε, ως ε, Προεδρία είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ ελπίζουμε να συνεργαστούμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για αντικειμενικούς λόγους. Είναι το θέμα της, του εξυγχρονισμού του νομικού καθεστώτος, κυρίως όσον αφορά τα συγγραφικά δικαιώματα. Αναφέρομαι τα δικαιώματα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το, τα δικαιώματα του δημιουργού και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ έθιξε το θέμα αυτό και είπε ότι ένα από τα πρώτα θέματα, θέματα πρώτης προτεραιότητας. Προτίθεται λοιπόν να καταθέσει νομοθετική πρόταση κατά τους πρώτους έξι μήνες από τότε που θα τεθεί σε ισχύ, που θα αρχίσει να δουλεύει, που θα αναλάβει τις δραστηριότητες της η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι οτι έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αλλά βέβαια να έχουμε καταρχήν κάποιες συγκεκριμένες εγγυήσεις, να έχουμε θετικές ε, διασφαλίσεις έτσι ώστε να μπορούμε στον τομέα αυτό να καταθέσουμε μία πρόταση η οποία θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση ε, της κοινωνικής αγοράς και κάτω από το ψηφιακό πρίσμα. Σήμερα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα δικαιώματα του δημιουργού και άλλα συναφή δικαιώματα και στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων αυτά τα δικαιώματα είναι εκτεθειμένα και γίνεται κατάχρηση αυτών λόγω ακριβώς της ψηφιακής εξέλιξης. Από την άλλη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα ε, που βασίζονται σε online διάδοση έργου αυτά έχουν πλέον συνεπάγονται και νέες εξελίξεις και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λιγάκι την κατανάλωση αυτών των θεμάτων. Είναι Ένα θέμα που χρήζει αντιμετώπισης και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αναθεώρηση του copyright, μια διαδικασία που προέκυψε από διαπραγματεύσεις με την σχετική επιτροπή. Βέβαια η επιτροπή είχε πει ότι θα υπάρξει λευκή βίβλωση επ' αυτού, τελικά δεν προέκυψε. Ε, θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει επ' αυτού ο κύριος Γιούνκερ. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε εγγυόμενοι την ισορροπία ανάμεσα στις νέες επιχειρήσεις, της νεοφυής ε, οι οποίες αποκαλούνται στον κοινωνικό τομέα αφενός και αφετέρου ισορροπία σας είπα με ένα νομοθετικό σύστημα το οποίο προσφέρει εγγυήσεις στα δικαιώματα του δημιουργού με προσαρμογές οι οποίες όμως ε, θα είναι ελάχιστες, δεν θα είναι τόσο σημαντικές, κυρίως όσον αφορά το σύστημα το οποίο ισχύει τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έχει φανεί έχει διαπιστωθεί ότι ισχύει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ισχύον σύστημα και για ψηφιακή χρήση. Όμως, όπως σας είπα, ε, με κάποια σύνεση διαφυλάσσοντας ε, τις ισορροπίες και διαφυλάσσοντας και τα συμφέροντα που διακυβεύονται. Θα δούμε τι θα προκύψει και από τις ε, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις της Επιτροπής. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα μου πείτε κύριε Πρόεδρε πόσα λεφτά έχω ακόμα, λεπτά έχω ακόμα για να συνεχίσω γιατί μήπως χρειάζεται να περάσουμε στις ερωτήσεις απαντήσεις αλλά τέλος πάντων ένα άλλο θέμα το οποίο ε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας ε, είναι οι εταιρείε περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο μέτοχο για μας ε, είναι θέμα προτεραιότητες για το λόγο που ανέφερα στην αρχή γιατί θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια στις διασυνορικές συνεργασίες και στον τομέα αυτό υπάρχει μια προφανής δυσκολία να λειτουργήσουμε σε διασυνοριακό επίπεδο λόγω ακριβώς της ανομοιογένειας ε, στις εθνικές νομοθεσίες και λόγω της έλλειψης ε, εμπιστοσύνης σε σχέση με τους πιθανούς πελάτες και σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ είναι μια κλασική περίπτωση όπου η αβεβαιότητα και ένα μη ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο εμποδίζει την πλήρη λειτουργία της οικονομίας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αφαίρεση εμποδίων ε, στις ε, διασυνοριακές συναλλαγές είναι για μας μια προτεραιότητα την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και στην ε, αναθεώρηση πολιτικής ε, για το, τη στρατηγική του 2020. Η, η Ιταλική Προεδρία ε, θα προτείνει μια οδηγία για, τα, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, δηλαδή εταιρείε περιορισμένη ευθύνη με έναν μέτοχο και θέλουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία ε, στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος του εξαμήνου ενδεχόμενα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαίρως και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ε, στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης. Υπάρχουν και άλλα θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Ένα να σας αναφέρω μόνο και ολοκληρώνω εδώ. Θα ακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ένα άλλο θέμα που είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις ε, εκτός αγροτικού τομέα. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε την, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κομισιό μέσα στα πλαίσια, μέσα στα πλαίσια της πράσινης βίβλου είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ε, τους Ευρωπαίους παραγωγούς ε, γιατί προστατεύει την παραγωγή τους και ε, περιορίζει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να διαθέσουν εμπορικά, να διαθέσουν στο εμπόριο τα προϊόντα τους εκτός της τοπικής αγοράς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες, ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε με με αποτελεσματικό τρόπο, διότι συνδέεται ε, και με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την εσωτερική αγορά. Και συνδέεται επίσης ε, και με τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματεύεται κάποια θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό πρέπει να επιληθεί με θετικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσει για την προώθηση και για την προστασία τη Ευρωπαϊκή παραγωγή και τη παραγωγή που έχει να κάνει με την, ε, με, τις, ε, με την ποικιλία αν θέλετε παραγωγής ε, στην, και την πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της ζήτησης ε, που θα λάβει η χώρα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 25ης Σεπτεμβρίου και θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Πολύ αρμόδια και πάρα πολύ ε, εύκολα αποδώσατε αυτά που ο υπουργό σα θα ήθελε να αποδώσει εδώ και να μας πει όσον αφορά τα θέματα τα οποία θα εξετάσετε και πραγματικά αυτό αγγίζει και τις καρδιές ακόμη των παρόντων εδώ σαν νομική επιτροπή και σαν πρόεδρος αυτής της επιτροπής θα ήμουν ευγνώμων ε, τις ανταλλαγές απόψεων που έχουν γίνει Ο κύριο Διρό είναι πρώτος. Ο κύριος Διρό. Παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Διρό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργό, Υπουργέ σα ευχαριστώ. Σα είχα ακούσει σε μια άλλη επιτροπή για τη χαρά αυτή. Μιλήσατε για το θέμα όσον αφορά τους πολίτες για τον κατάλογο των λόμπι ενδιαφέρομαι εγώ πάρα πολύ για αυτό το θέμα αλλά είμαι ανήσυχο παράλληλα για ένα θέμα το οποίο συνάπτεται όσον αφορά το εμπιστευτικότητα της, των business. Αναφερθήκα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα πρέπει να προσεγγίσει την αμερικανική νομοθεσία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η του Συμβουλίου αλλά και την αίσθηση την οποία έχετε εσύ, εσείς όσον αφορά την ισορροπία μπορούμε να βρούμε μεταξύ προστασίας της οικονομικής δραστηριότητας η οποία προστατεύεται από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά την πνευματική ε, ιδιοκτησία, την προστασία από τον ανταγωνισμό, αθέμητο, τον ανταγωνισμό, με, δεν, δεν υπάρχει κανένας ορισμός πράγμα το οποίο δεν, είναι, δεν συνάδει με το δίκαιο το παραδοσιακό που είναι διαφορετικό του αγγλοσαξονικού. Κατά αυτόν τον τρόπο λέγω, όσον αφορά το εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών, μήπως δεν, κατά αυτόν τον τρόπο θα εμποδίσετε ορισμένε πληροφορίε, διότι υπάρχουν πληροφορίε που είναι παράνομα τις συλλαμβάνουν μερικοί. Και είμαι πάρα πολύ ανησυχικό εγώ σε σχέση όταν αφορά τη διαφάνεια, ό,τι αφορά οποιοδήποτε συναγερμό που έχει γίνει για μη κανονικές συμπεριφορές των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τους παραδείσους, ε, φορολογικούς παραδείσους κλπ. Και αυτά τα θέματα είναι μείζωνα για την ψηλονέψηνα και για τους πολίτες μας. Αλλά για παρά πληροφορία περνάει από την προστασία μέσα από τους δημοσιογράφους, μέσα από το συνογερμό, καθώς μέσα από αυτούς οι οποίοι καταγγέλνουν τέτοια πράγματα, πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ βαριά θα έλεγα. Κατά πόσο πραγματικά εσείς κύριε Υπουργέ θα προσπαθήσετε να έχετε μια ισορροπία όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο επόμενο αγορητή, κύριε Χακνέρ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ για τις τόσες πολλές πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω ότι η Ιταλική Προεδρία ε, φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Ε, μίλησατε για ένα σωρό θέματα, για τα εμπορικά σήματα, για τα εμπορικά μυστικά και πάρα πολλά άλλα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα εμπορικά μυστικά, τα trade secrets. Ε, και εγώ θέλω να πω το εξή Πολύ συχνά βλέπουμε ότι επιχειρηματικά μυστικά αυτό πολλές φορές λέγεται για να αποκρύψουν οι επιχειρηματίες ε, πληροφορίες από τους εργαζόμενους και από τα επιχειρησιακά συμβούλια. Τους ε, λένε και ισχυρίζονται ότι πρόκειται για επιχειρηματικό και ε, εμπορικό μυστικό ε, για να αποφύγουν του εργαζόμενους. Έτσι λοιπόν η Ιταλική Προεδρία τι προτείνεται να κάνει, πώς θα μπορέσει ε, να συμπεριλάβει τους εργαζόμενους αυτούς και σε συζητήσεις που μέχρι τώρα δεν συμμετείχαν. Και μία άλλη ερώτηση που θα είμαι λίγο κουραστική γιατί έκανα την ίδια ερώτηση και στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ στην ε, δική μας την Επιτροπή δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα Υπουργεία μιλήσατε πολύ ε, για την εταιρική governance. Μιλήσατε για τις γυναίκες στα εποπτικά συμβούλια. Έχουμε ψηφίσει επ' αυτού του θέματος και τώρα ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης μας έδωσε κάποιες πληροφορίε, αλλά νομίζω ότι εσείς θα είσαστε περισσότερο αρμόδιος και γι' αυτό μας ενδιαφέρει τι προτίθεται να κάνει η Ιταλική Προεδρία, όχι έτσι γενικά και αόριστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα στις ομάδες εργασίας. Το επόμενο θέμα που θέλω να, θέξω, να θίξω αφορά στην ανταγωνιστικότητα. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας ε, το παρουσιάσατε κάτω από διάφορα οπτικά πρίσματα ε, το τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, εγώ είμαι μία εξ αυτών που είναι κράτανε τα πεπισμένη ότι την ανταγωνιστικότητα πρέπει να την εξετάζουμε στο πλαίσιο ενός τριγώνου. Βεβαίως και πρέπει να είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό προς τα κάτω. Κάθε άλλο θα πρέπει να διαφυλάσσονται παράλληλα και τα συμφέροντα και των εργαζόμενων αλλά και των ε, καταναλωτών. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν ε, αρκετές ε, υπερβολές, ε, τις είδαμε αυτές τις υπερβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τώρα πλέον θα πρέπει να προβούμε σε λήψη κάποιων συγκεκριμένων μέτρων και μέσω της governance. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν θεσπιστεί και έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς Πρόκειται για αυτήν την ε, μίνι ΕΠΕ που την παρουσιάσατε. Η Ιταλική Προεδρία τι προτίθεται να κάνει πολύ συγκεκριμένα έτσι ώστε να προάγει το θέμα αυτό. Και αυτό πάντα κάτω από το πρίσμα ότι θα πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων, των καταναλωτών, γενικά τα δικαιώματα των πολιτών και όχι να επιδιώκει τον ε, ανταγωνισμό που οδηγεί πάντα σε ολισθηρό δρόμο προς τα κάτω. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, <laughs> κύριε Υπουργέ. Ήταν πλήρη ο λόγο σα όσον αφορά τι προτεραιότητε τη Τελική Προεδρία. Ένα θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι το σημάτο και τα πρώτα βήματα τα οποία είχαμε σαν αφορά μια συμφωνία που έχει γίνει στο επίπεδο του Συμβουλίου σαν αφορά τα σήματα. Φρονώ πως η εργασία η οποία θα πρέπει να γίνει μεταξύ αυτών των διαφόρων οργάνων, κομισιών, κοινοβουλίου κλπ. Αλλά θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα εξή σημεία, δύο σημεία συγκεκριμένα. Φαίνεται πως η πρόταση του Συμβουλίου είναι όσον αφορά τον έλεγχο των εμπορευμάτων που είναι σε transit, ποιοι είναι οι όροι, ποιοι, τι επελέγησαν σαν κριτήρια όσον αφορά αυτόν τον έλεγχο και δεύτερο σημείο, ποιοι τρόποι υπάρχουν για τη συνεργασία των OSMI, το ευρωπαϊκό, και τους εθνικό ε, ομάδες των ευρωστοχνιών και σημάτων. Είναι στοιχεία τα οποία αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπάρχουν πτυχές τις οποίες πραγματικά θα ήθελα να μας διευκρινίσετε. Ένα άλλο θέμα είναι όσον αφορά τα συγγραφικά δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα. Επεξηγήσατε πώς η αναταραχή η οποία έχει λόγω του των νέων συστημάτων και πώς αυτά εφαρμόζονται στα νέο οικονομικό μοντέλο. Σε αυτή την αναταραχή λοιπόν η εργασία η οποία θα πρέπει να έχει επιτελεστεί είναι η εργασία αλλά φρονώ πως πρέπει να επακρυπνούμε γιατί βλέπουμε πως πραγματικά έχουμε μια αναταραχή και μια ανατροπή των πραγμάτων με την ανάκυψη των αυτών των νέων επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία, με αυτά τα νέα τεχνολογικά των ψηφιακών εργαλείων και οργάνων αν θέλετε και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να μας διασφαλίσετε ότι τα ποσά τα οποία συγκεντρώνουν θα πηγαίνουν προς τους δημιουργούς, τους, τα πνευματικά δικαιώματα, τα copyright κλπ. Και κάτι ακόμη το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως είναι το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Όντως είναι ένας τρόπος για να υπάρξει μια αξιοποίηση ενάντια σε αυτή τη ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στην υπερβολική για να μπορεί να εξασφαλιστεί μια εργασία η οποία θα είναι τοπική και η οποία αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα θα μπορεί να βοηθήσει στην πρόθεση των προγραμμάτων αυτών, των, συγγνώμη, των επιχειρήσεων αυτών προς τα έξω, προ τις τρίτε χώρες εκτός κοινότητα και κατά πόσο η Κομισιόν αυτή τη στιγμή συνάδει με αυτή την άποψη και κατά πόσο είναι μια πρόταση η οποία, στην οποία συγκατατίθεστε κι εσείς ούτως ώστε να καταταθεί ενώπιον του Συμβουλίου την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έσχατος ο κύριος Καβαντά παρακαλώ. Πάμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, πρόεδρε. Αγαπητέ Σάντρο. Είστε βουλευτής και ε, παλαιότερα μπορούσαμε να μιλάμε και μάλιστα σας μιλούσα στον ελληνικό. Σας θυμάμαι εδώ και θα πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τώρα που σας μιλάω κύριε Υπουργέ αλλά ωστόσο ένας βουλευτής ο οποίος άσκησε για πολλά χρόνια τα καθήκοντά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν έρθει στην εξουσία είναι κάτι σημαντικό. Σας λυπάμαι γιατί το εξάμεινο της τελική Προεδρίας έχει τέσσερις μήνες, είναι τετράμινο. Θα χαρώ όμως αφετέρου, αλλά Ιούλιο και Αύγουστο, ξέρω εσείς δεν καθίσατε, δεν οκνηρείτε ε, προετοιμάσατε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τους προσανατολισμούς, τις εργασίες για μια νέο ξεκίνημα της Ευρώπης καθότι το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα έκτακτο λόγω του σκεπτικισμού που εμφανίστηκε σε ευρωπαϊκές εκλογές αλλά επίσης και αυτή τη νέα, το νέο τοπίο το οποίο έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πραγματικά οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν γεράσει περισσότερο. Αυτή η προεδρία λοιπόν Ιταλική, το είπα προηγουμένω και το είπα και στον συνάδελφο στον κύριο Ρολάντο, είναι κάτι σημαντικό καθότου, διότι αν τα λόγια ακολουθούν, τις πράξεις ακολουθούν τους λόγους, ο οποίος, αν πρωθυπουργός της Ιταλίας, μπορεί κάλλιστα να δώσει νέα πνοή στην Ευρώπη διότι η κρίση δεν κτύψε μόνο τη χώρα σας αλλά και δεν είναι μόνο η χώρα αλλά θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα εμψύχωση των πολιτών ότι ασχολούμεθα με τα ουσιώδη θέματα και όχι τα επουσιώδη. Και αυτό υπήρξε το σημείο το οποίο υπογραμμίσατε. Ένα άλλο σημείο για το οποίο θέλω να επιμείνω αγαπητέ Σάντρο είναι ότι η αίτησή μου είναι ότι μια, μια η οποία πραγματικά κάνει μια προσπάθεια για να λειτουργήσει και ότι αυτή τη στιγμή επειδή έχω την περηφάνεια να ασχοληθώ με αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα ότι δεν είναι κλειστή μια επιπυρός αλλά ότι είναι ανοιχτή Μία αρχή είναι αυτή η οποία πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανά να εφαρμόσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά την υπηκορικότητα για την ευρωπαϊκή επικοδόμηση. Αυτό είναι το γενικό κάδρο. Όταν εσείς προηγουμένως είπατε ότι υπάρχει πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και να προσθέσω, το πρώτο είναι ότι ασπάζουμε την άποψή σας και λυπάμαι αυτή την άποψη ότι, ότι η Προεδρία σας δεν ξεκαθάρισε αυτή την κακή συνήθεια που υπάρχει ότι τα ελάχιστα, τα, τα κείμενα τα οποία είναι ελαχίστης ε, σημασίας αποτελούν ευρωπαϊκή πολιτική αυτόματη φημή προς τα έξω. Πιστεύω ήταν στο πρόγραμμά σας να κάνετε την πολιτική με την ευγενή μορφή της πολιτικής και όχι να γίνει μια τεχνοκρατική πολιτική η οποία είναι η πολιτική της νομοθέτησης των ευρωπαϊκών νόμων και νομίζω πως αυτό θα είναι υπέρ των ευρωπαϊκών λαών και πιστεύω πως πρέπει να διατηρηθούμε τι χρησιμεύει το δίκαιο σε αυτή την Ευρώπη. Και ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η δύναμη της Ευρώπης εγκρίνω το ενδιαφέρον το οποίο έχετε ημών ε, σου σάντρο του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης και του Πρωθυπουργού σας όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Δείτε, δύο ε, πύρους, Ευρώπη, Αμερική, βλέπουμε δύο πράγματα διαφορετικά. Αυτοί οι οποίοι προμηθεύουν τα πράγματα και προμηθεύουν την ευρωπαϊκή ιδέα κατά μεγάλο βαθμό. Δύο τρίτα προ ένα τρίτο σε ό,τι άπτεται ε, την παραγωγή, την παγκόσμια παραγωγή. Πολλοί φρονούν ότι δεν είναι απαγορευμένο να, να κλέψουν κάτι και ότι η πάση μπορεί να κλέψει ό,τι θέλει οποιοδήποτε έργο. Εσείς είπατε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κουλτούρα, πολιτισμός χωρίς μια οικονομία της κουλτούρας και βεβαίως όσον αφορά τα δικαιώματα, τα συγγραφικά, τα πνευματικά δικαιώματα. Ε, αυτά τώρα εδώ και πιστεύω θα με καλέσετε για ένα καφέ και θα με ξεχάσετε. Κύριε Υφυπουργέ, δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κατάλογο, γι' αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω να πάρετε το λόγο και να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ξεκινήσω απαντώντας την τελευταία παρέμβαση και να χαιρετήσω τον κύριο Ζωμαρή Καβαντά, τον αγαπητό φίλο Ζωμαρή και να απαντήσω στα θέματα τα οποία έθιξε. Δεν αναφέρθηκα ρητά σε αυτό στο θέμα της επικουρικότητας. Αλλά πολύ καλά κάνατε, κύριε Καβαντά, που το θίξατε. Είναι ε, ε, αυτονόητο, διότι από τη μία πλευρά, όπως είπατε και μας ενθαρρύνατε Κοιτάξτε, τρία χρόνια στην Προεδρία, αυτό είναι απειλή για την υγεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο, αλλά δεν χρειάζεται. Και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, η επικουρικότητα είναι αυτονόητη, διότι όταν έλεγα ότι χρειάζεται να ε, καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατική υπερβολή. Εμείς στην χώρα μου είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις ε, υπερβολές της γραφειοκρατίας Δημοκρατίας και μιλάμε για την αντίστροφη ε, ε, γραφειοκρατία, ε, αντίστροφη συγγνώμη, επικου, επικουρικότητα, είναι ένα θέμα ας πούμε ένα, για παράδειγμα το ελαιόλαδο Υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός στον τρόπο με τον αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ελαιόλαδο. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή ε, παραγωγή σε διεθνές ε, επίπεδο και ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής γίνεται μέσω των εμπορικών συμφωνιών και όμως οι παραγωγοί μας ε, στην χώρα μου παραδείγματος χάρη θεωρούν ότι δεν γίνεται καλά η δουλειά στην, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως ε, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο να πούμε θα σερβίρουν το λάδι στο τραπέζι η Ευρώπη δεν πρέπει να μπαίνει σε τέτοιου είδου λεπτομέρειες και να προσπαθεί να διδάξει στους ταλούς πώ θα σερβίρουν το λάδι. Αντίθετα, θα πρέπει να κάνει μια δουλειά υπέρ των παραγωγών, να διασφαλίσει δηλαδή, τα συμφέροντα των παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο διεθνές ευώριο. Εμείς ξεκινήσαμε και συνεχίσαμε μάλλον το έργο της ε, ελληνικής προεδρίας, το διευρύναμε το συζητήσαμε και στο άτυπο συμβούλιο του Μιλάνο και θεωρούμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην έναρξη της νομοθεσίας και στην έναρξη αυτού του νέου πολιτικού κύκλου πρέπει να σκεφτούμε πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς λειτουργήσε ε, συγκεκριμένα και όχι μόνο στα θέματα επικουρικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, ε, λειτουργία της γιατί πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις αρχές το πλαίσιο και μετά να μπούμε σε λεπτομέρειες. Και αυτό το πλαίσιο σχετίζεται με τη λειτουργία και του Συμβουλίου ΜΕΝ, των Υποσυμβουλίων Υπουργών, αλλά και με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι ε, όλες οι προεδρίες ε, έχουν αναλάβει τη δέσμευση να υποβάλουν μία ε, έκθεση για τον τρόπο αυτών λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την διαθεσμική συνεργασία, για τα θέματα επικουρικότητας και τα θέματα αναλογικότητας και φαίνεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος ο κύριος Γιούνκερ έχει κάποιες ε, καθησυχαστικές ε, προτάσεις ε, για το μέλλον και θέλει να εστιάσει την προσοχή του περισσότερο στον πυρήνα, στο core business της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό οι προεδρίες θα το ενθαρρύνουν. Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της δημιουργικότητας και της πνευματικής ιδιοκτησίας και των νέων τεχνολογιών. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά, ε, σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καβαντά και ο κύριος Ροζιέ, διότι αναφερθήκατε σε μια προτεραιότητα την οποία έθιξα και εγώ που μας απασχολεί άμεσα είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, αυτό το, αυτή τη δημιουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, να προστατεύσουμε τους δημιουργούς, αυτούς που παράγουν πολιτιστικό έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προωθήσουμε επίσης την τεχνολογική εξέλιξη. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε την, την εξέλιξη, την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύσουμε τη δημιουργικότητα και την τέχνη. Και εμείς έχουμε πρόθεση, την πρόθεση να συνεργαστούμε ακριβώς όπως είπατε και εσείς. Στο θέμα των εμπορευμάτων που βρίσκεται σε transit ε, σε αυτό που είπατε για το trade package στα θέματα των, του ελέγχου αυτών των εμπορευμάτων πρέπει καταρχάς να σεβαστούμε τους διεθνείς κανόνες Είπατε ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την νομικότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα νόμιμη αυτή η έλεγχη. Αλλά μετά και μετά την ε, μια δύσκολη συζήτηση, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου επιβεβαίωσε τη θέση αυτή και θεωρούμε ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη και ισορροπημένη θέση την οποία να έχουμε πετύχει όσον αφορά τα παραχαραγμένα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε τράνζιτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα ε, ε, εμπορεύματα αποτελούν ε, ένα μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη του εμπορίου, για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών και των καταναλωτών. Όλοι αυτά είναι λόγοι για να υπερασπιστούμε αυτή την συμφωνία που είναι πάρα πολύ δύσκολη και την οποία πετύχαμε σε, επίπεδο του Συμβουλίου. Είναι μια συμβιβαστική λύση αυτή. Είναι όμως μια θέση η οποία μας ικανοποιεί. Δύσκολα την πετύχαμε, αλλά εάν ανοίξουμε ένα κάποιο σημείο τώρα της συμφωνίας αυτής, κινδυνεύει να καταρρεύσει όλη η συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τις ε, επιχειρήσεις με έναν μέντοχο και του corporate governments. Ε, αναφερθήκατε στο θέμα της ε, συνδιαχείρισης. Ε, όντως υπάρχει μια ρήτρα διασφάλιση, μια ρήτρα ασφάλειας για την συνδιαχείριση στην οποία αναφερθήκατε και πιστεύουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανησυχιών που εκφράσατε, θεμητών ανησυχιών μεν, ε, επιλύονται από αυτή την ρήτρα διασφάλισης. Τώρα, για το άλλο θέμα το οποίο αφορά τις δύο βασικές ελευθερίες τις οποίες έθιξα στην αρχή της παρέμβασής μου γιατί είπα ότι το εξάμεινο αυτό θα έχουμε κάποιες βασικές προτεραιότητες ε, κάποια θέματα φάρους που είναι παραδείγματος η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της ενημέρωσης η ελευθερία ε, της ε, ενημέρωσης των καταναλωτών. Αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά και σκεφτήκαμε ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφεύγουν ε, αυτή τη στιγμή στο εμπορικό απόρριτο διότι δεν έχουν τα μέσα, τους, τους χρηματικούς πόρους για να καταχωρήσουν τα σήματά τους, τα, να καταχωρήσουν τα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να τις προστατεύσουμε μεν, αλλά να μην περιορίσουμε και ε, υπερβολικά το δικαίωμα ενημέρωσης, το οποίο πολύ σωστά αναφέρατε. Τώρα, για τις... Ε, Ε, ε, κάτι ένα θέμα το ποσοστό σου που έδειξε η κυρία Ρέγνερ. Εμείς ε, σαν Ιταλοί έχουμε την καλύτερη εμπειρία. Το, οι ποσοστώσεις για την, παρουσία, για την παρουσία των δύο φίλων στις επιχειρήσεις. Εμείς ξεκινήσαμε από το 16%, τώρα έχουμε 30% ε, στην Ιταλία. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά η νομοθεσία μας σε, Ευρώπα, σε ιταλικό επίπεδο, αλλά δεν ε, ε, βλέπουμε γιατί να μην λειτουργήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φιλοδοξία μας είναι βέβαια να έχουμε ένα γενικότερο προσανατολισμό στο Συμβούλιο. Ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μειοψηφία που μπλοκάρει τις εξελίξεις και προσπαθούμε να πετύχουμε μια ειδική πλειοψηφία, δηλαδή να πείσουμε κάποιες χώρες και ίσως ακόμα και εσείς θα μπορούσατε να τίνετε μια χείρα βοηθείας, θα μπορούσατε να πείσετε κάποιες χώρες ε, για να βγούμε από το αδιέξοδο ε, και να καταλήξουμε σε μια ε, πιθανή λύση δηλαδή να βρεθεί μια δυνατότητα να πάρουμε μια απόφαση. Τέλο πάντων, εμείς θα καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια για να για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό των ποσοστώσεων ε, εκπροσώπησης και των δύο φύλων. Είναι προ όφελό μα στην Ευρώπη. Εμεί στην Ιταλία είχαμε μια καλή εμπειρία μέχρι στιγμή. Και νομίζω. Α, όχι, όχι, να αναπίνησα. Ε, ε, θίξατε επίση και το των μη, γεω, των μη, αγροτικών ε, γεωγραφικών ε, προσδιορισμών. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που κατά την άποψή μου παίζουμε την εμπιστοσύνη ε, ανάμεσα στην Ευρώπη και στους ε, Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως ανάμεσα στην Ευρώπη και στους μικρούς παραγωγούς και θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι να διδαχθούν από τα διδάγματα του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος συγκεκριμένα να υιοθετήσουμε δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση αλλά και πιο συνεκτική ε, αντιμετώπιση και όσον αφορά τα, κυρίως τα βιομηχανικά μας συμφέροντα διότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ε, τους παραγωγούς, τους μικρούς παραγωγούς, τους παραγωγούς ε, παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων διότι θα πρέπει να ε, προωθήσουμε αν θέλετε τις ε, παραγωγές τις τοπικές ε, που έχουν να κάνουν και με την πολιτιστική παράδοση μιλάμε για γενικότερες παραδόσεις που θα πρέπει να διατηρηθούν και εδώ αναφέρομαι και στην επικουρκότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, και εδώ είναι προφανής η περίπτωση, εδώ χρειάζεται και μία ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προστασία των καταναλωτών, προστασία των δικαιωμάτων. Δηλαδή χρειαζόμαστε και επαναλαμβάνω μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους οικονομικούς λόγους που ανέφερα αλλά και γιατί σήμερα υπάρχουν δυσκολίες ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες οι παραγωγοί για να διαθέσουν στο εμπόριο τα προϊόντα τους εκτός ε, της περιοχής τους διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει η νομοθεσία μας ε, να αναπτυχθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και είναι προφανές ότι από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να ε, ρυθμίσουμε σε νομικό επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο, συγγνώμη, ε, να εναρμονίσουμε ενδεχόμενα και τις πολιτικές μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα των γεωγραφικών προσδιορισμών, αλλά αυτό θα εξαιρεθεί από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε εμείς το θέμα, από τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούμε εμείς στις διάφορες εμπορικές διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε με τις τρίτες χώρες. Υπάρχει μια άμεση σχέση και όσον αφορά την νομοθεσία αλλά και την θέση, την πολιτική θέση ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο εμείς στο εσωτερικό επίπεδο θα ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά και στις ε, διεθνείς μας ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε σκληρά. Θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, τέλος Σεπτεμβρίου και έτσι όπως σας μίλησα εγώ σήμερα θα το θέσουμε και στο Συμβούλιο ενώπιον των Υπουργών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Mr. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υφυπουργέ που κατορθώσατε το ακατόρθωτο να καλύψετε τόσο σημαντικά θέματα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι η Επιτροπή αυτή ε, περιμένει πάρα πολλά από την Ιταλική Προεδρία και είμαι σίγουρος ότι στο πρόσωπό σας ε, θεωρούμε ότι είστε ο άνθρωπος που θα βοηθήσει να επιτύχουμε πάρα πολλά κατά τους επόμενους έξι μήνες. Σας ευχαριστούμε.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 If you kindly permit me, I will continue the meeting. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Ησυχάστε παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ για την ησυχία. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προεδρείου. Εξή. Ο Τζόναθον Φολ, Γενικό Διευθυντή τη Γενική Γενική Διεύθυνση Ιστορική Αγορά, καλεί τα μέλη τη Επιτροπή να παρακολουθήσουν μια συ... συνέντευξη που θα γίνει αύριο 4 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αναφορά την καινοτομία Δεδομένη τη αρμοδιότητα τη Επιτροπή αυτή για τα θέματα αυτά, νομίζω πω θα είναι τεράστια σημασία σε αυτή, αυτό το συνέδριο για όλου εδώ του βουλευτέ, καθώ επίση, αν θέλετε, η Γραμματεία μπορεί να σα δώσει περαιτέρω πληροφορίε για αυτή τη συνάντηση. Τα μέλη λοιπόν καλούνται στην δεξίωση που θα γίνει υποδοχής στις 6.30 θα γίνει ενώπιον αυτής της έξω από αυτή την αίθουσα το καλωσόρισμα. Μια άλλη ανακοίνωση είναι ότι έχουμε μια απόφαση η οποία διευθυνθεί από τους συντονιστές σήμερα το πρωί εάν συμφωνείτε η γραμματεία θα το κυκλοφορήσει γραπτός αυτά τα οποία αποφασίστηκαν και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Είμαι εισηγητές των διαφόρων εκθέσεων και Θέλετε να περάσω όλα τα σημεία αυτά ένα προς ένα σε αυτή τη συνεδρίαση. Παρακαλώ κυρία Γιάννη, παρακαλώ, έχετε λόγο. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μας τα δώσετε σε γραπτή μορφή, γιατί πρόκειται για μια συνάντηση των συντονιστών ε, που ήταν ε, ιδιαίτερα διεξοδική, αλλά απλά να πω έτσι κανονικά, ε, σε άλλη περίπτωση, όλα αυτά λέγονται και προφορικά. It's in writing. Α, μικροφόνο πρόεδρο. Α, ζήτησαν, μπορεί να τα δώσει γραπτό, Μάλιστα, συμφωνούμε, λαμπρά. Σημείο 3. Πρακτικά τη προηγούμενη συνεδρίαση. η συντακτική τη 7 η Ιουλίου και την έκτακτη τη 10 η Ιουλίου ενεστώτησέ του. Υπάρχουν αντιρρήσει όσον αφορά την έγκριση των πρακτικών, ουχή, λαμπρά, υιοθετούνται. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο σημείο 7. Δεν, δεν κάνω λάθο λοιπόν. Είναι θέμα το οποίο επανέρχεται είναι από τη Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τι δραστηριότητε και επιβλίωση και επίβλεψη των θεσμικών οργάνων για, την, για τις διατάξεις που έχουν σχέση με την συνταξιοδότηση. Ξέρετε, έρχεται εκ μέρου τη νομική επιτροπή, νομική υπηρεσία και αυτοί συμφέρανε πω αυτή η πρόταση δεν δημιουργεί νέα τροπολογία οποιαδήποτε και η γραμματεία της Επιτροπής μας συμφωνεί ότι προτείνει όπως η Επιτροπή αυτή υιοθετήσει την άποψη αυτή ως έχει υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα λαμπρά ουχή δεν βλέπω αντιρρήσει, αλλά θα το θέσω σε ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ αυτή τη προτάσεω τη νομική υπηρεσία, βεβαίω. Κατά. Αποχέ. Λαμπρά. Το σημείο 8 έχει αναβληθεί όσον αφορά τον ο κώδικα για τις βίζες τώρα επί την επικορικότητα σημείων 9 Έχουμε μία άποψη από το Λευθερονικό Κοινοπούλιο από το θέμα. Μπορώ να ζητήσω την κυρία Τελβόρ, σαν την κυρία Τελβό, να κάνει μερικέ παρατηρήσει, οι οποίε θα ήθελα επί του αυτού. Κυρία Τελβό, έχετε Έχουμε δεκτή συνουσία δύο Και ε, δεν είναι μόνο η Σουηδική, αλλά είναι και η Σουηδική, το Σουηδικό Κοινοβούλιο το οποίο μας έστειλε, οι οποίοι αντούν τη νομική βάση. Το θέμα είναι τη νομική υποδομή όσον αφορά τι εχειρώσεις που μπορεί να υπάρξουν εναντίον των πολιτών. Το άρθρο 36 προβλέπει τέτοια μέτρα για τα τη μελη αλλά αν δεν προβλέπει ο, τον κατάλογο των κυρώσεων που θα πρέπει να υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δούμε το άρθρο 83. Αλλά ξέρετε αυτό το άρθρο είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω μια τάση να ακολουθήσω την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας αυτής. Ξέρετε το θέμα αυτό των τελωνίων και της παραβιάσεων είναι κάτι το οποίο είναι κοινό. Μήπως η νομική υπηρεσία έχει κάτι άλλο να προσθέσει, κάτι άλλο να πει. Ασχόλιο, σχόλιο, παρατηρήσεις. Νομική υπηρεσία έχει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ναι, πρόεδρε. Όχι, δεν θα είχα τίποτα να προσθέσω πέρα από αυτές τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί και είναι οι θέσεις μας. Ευχαριστώ. Μπορούμε να έρθουμε στο επόμενο σημείο. Αναβάλαμε. Το σημείο 10 επίσης ανεβλήθη. Τα επόμενα σημεία και κλεισμένο των θυρών θα παρακολούσα λοιπόν αυτού οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην αίθουσα αυτή να εγκαταλείψουν στην αίθουσα παρακαλώ διότι η συνεδρία θα συνεχιστεί και κλεισμένων των θυρών.